Όθηση τη επιχειρηματικότητα των νέων μέσω τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση. Η συγγήτρια έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή στην έκθεσή μου. Πρόθεση τη επιχειρηματικότητα των νέων μέσω τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση. Ξέρετε ότι προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε πάρα πολλές γνώσεις κατά τη σύνταξη της έκθεσης αυτής και θεωρώ ότι καταλήξαμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Οι επιχειρηματικές δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν, μπορούν να αποκτηθούν και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την κοινωνία. 225 είναι τροπολογίε οι οποίε υποβλήθηκαν για την έκθεση αυτή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι ενδιαφέρονται για αυτή την έκθεση και πρέπει να πω ότι συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά με του κοιόδη ηγητέ από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω τη έκθεση αυτή προσπαθεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα τη υψηλή ενεργεία των νέων που φτάνει το 50% σε κάποιε χώρε. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων Ωστόσο, αυτή είναι η μόνη έκθεση η οποία έχει υποβληθεί για το ζήτημα αυτό. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει οι νέοι να μπορούν να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δεξιότητες και ότι ε, θα πρέπει να είναι σε θέση μέσω των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, είτε είναι τυπικά, μη τυπικά ή άτυπα, να μπορούν να αποκτούν επιχειρηματικές δεξιότητες. Στην έκθεση προσπαθούμε να καθορίσουμε αυτές τις επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες, καθώς επίσης και τα προγράμματα κατάρτισης που θα μπορούσαν να διδάξουν αυτές οι ικανότητες στους νέους. Λέμε ότι ε, θα πρέπει να προωθηθούν τέτοια προγράμματα τα οποία θα πρέπει να έχουν ε, μια διάσταση διαβίου μάθησης και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε την καινοτομία και τη δημιουργικότητα των νέων. Νέοι οι οποίοι θα είναι σε θέση να αναλάβουν κινδύνους και να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις. Η πρόκληση αυτή είναι τεράστια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε εδώ πέρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας δείξει προτραστική στάση μας έχει ήδη δώσει κάποια δεδομένα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus Plus από την περίοδο 2020 και μετά έχει αποφασίσει να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα των νέων και συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης των νέων όσον αφορά το επιχειρηματικό πνεύμα. Ήδη όμως από το 2016 πρόκειται να δοθούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια έκθεση για τις βέλτισες πρακτικές σε αυτόν τον τομέα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει όμως να περιμένουν την έκθεση αυτή, θα πρέπει από τώρα να αρχίσουν να προωθούν την επιχειρηματικότητα των νέων. Μολονότι αυτή αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο συστηματική ούτε τόσο καλά συντονισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να προτείνει μέσω τη έκθεση αυτή συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη, μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τι νεοσύστατε επιχειρήσει. Και όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γενικά προγράμματα για την προώθηση τη επιχειρηματικότητα και τη απασχόληση των νέων, όπω σα είπα το πρόγραμμα Erasmus Plus και το καθεξής. Οι διδάσκοντε επίση διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο κάνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη να αρχίσουν τώρα να προετοιμάζουν την ίδια την κατάρτιση των διδασκόντων. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η προώθηση τη επιχειρηματικότητα των νέων θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία και γι' αυτό το λόγο ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει στο μέλλον μια έκθεση προόδου όσον αφορά την πρόοδο που θα έχουμε επιτύχει. Σα ευχαριστώ πολύ για τη θετική σα συνεργασία και θέλω να ελπίζω ότι τα μέτρα τα οποία προτείνουμε στην έκθεση αυτή όντω θα προωθήσουν και θα βελτιώσουν την ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτιση και εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα των νέων. Νομίζουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε ευρύτερα και την κοινωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now for, for one minute, please. Mr. Venta. Ένα λεπτό, κύριος Βέντα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια. Πολύ σημαντικά θέματα της απασχόλησης των νέων θίγονται και καλύπτονται εδώ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα εξή. Η κοινωνική οικονομία και η υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας είναι σημαντική υπόθεση, ιδιαίτερα για τους νέους. Τέτοιες επιχειρήσεις όχι μόνο μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις να ανακάμψει η οικονομία, αλλά και συνεισφέρουν η κοινωνία συνολικά να μπορέσει να μετεξελιχθεί. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν, επιθυμούν η εργασία τους όχι μόνο να είναι αποτέλεσμα κάποιας ε, προτίμησης ή επιλογής αλλά να μπορούν επίσης να καλύπτουν και τις οικονομικές τους ανάγκες και να δημιουργήσουν και ίδιο κεφάλαιο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι νέοι να τύχουν κατάρτισης και εκπαίδευσης όσον αφορά ειδικά την εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση. Γι' αυτό χαιρετίζουμε την έκθεση. Κυρία Κώστα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ και ο Επίτροπος, γιατί πραγματικά πρέπει να αναλάβει τη σημαντικότητα αυτή δέσμευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ευχαριστήσω την συνάδελφο για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και νομίζω ότι το να λέμε ή να πρέπει να συνεχίσουμε να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες, ιδίως ανάμεσα στους νέους και είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προσανατολίσουμε τον κατάλληλο τρόπο τα εκπαιδευτικά σχολικά προγράμματα αλλά και τα πανεπιστημιακά προγράμματα για μια προώθηση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας και ενός επιχειρηματικού πνεύματος. Νομίζω ότι όπως υπόθηκε θα πρέπει να προωθήσουμε μέσω των προγραμμάτων αυτών και την απασχόληση. Ένα στου δύο νέου αυτή τη στιγμή μα λένε ότι στο μέλλον θα ήθελαν να κινηθούν αυτόνομα όσον αφορά την επαγγελματική του σταδιοδρομία και να δημιουργήσουν τη δική του επιχείρηση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρουμε να συνοδεύσουμε αυτού του νέου πολίτε. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προσφέρουμε στου νέου αυτού τα κατάλληλα προγράμματα κατάρτιση, αλλά κατάλληλα προγράμματα κατάρτιση των δασκόντων. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κύριο Σχέτμαν ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πέρσι στο Λουμπλίν παρακολούθησα, είχα διοργανώσει μια διάσκεψη νέων, ένα συνέδριο, ώστε να μπορέσουν να ενθαρρυνθούν, να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Με συζητήσεις με αυτούς τους νέους κατέληξα στο συμπέρασμα ότι τα εμπόδια τα οποία υφίστανται έχουν τον εξής χαρακτήρα. Δηλαδή, εκείνο το οποίο απουσιάζει είναι οι ιδέες ή το επιχειρήν, οι ιδέες για το επιχειρήν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να υλοποιηθούν οι ιδέες τους και να ε, υπερβούν τις δυσκολίες. Χρειαζόμαστε μια εκστατεία ενημέρωσης. Πώς για παράδειγμα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα κονδύλια που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν για, την, ε, για το επιχειρήν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ορισμένε από τι προκλήσει ε, που βλέπουμε είναι κοινέ ε, για όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλε πάλι δεν είναι κοινέ. Ε, υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στα κράτη-μέλη και θα ήθελα να μιλήσω για την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί πραγματικά έχουμε ένα πολύ ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα, όμω συχνά ακολουθούμε λάθο κατεύθυνση. Εκπαιδεύουμε σε λάθο τομεί. Του πιέζουμε σχεδόν το ίμιση των φοιτητών να πάνε στο πανεπιστήμιο, όμως δεν υπάρχουν τόσες ε, πολλές ε, θέσεις ε, και για να καταληφθούν στη συνέχεια χρειαζόμαστε επιχειρηματικότητα, κατάλληλη εκπαίδευση ούτως ώστε να τους κατευθύνουμε αυτούς τους νέους. καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης να μην παρεμποδιστεί ελεύθερη κυκλοφορία και βλέπουμε ότι ορισμένα μέτρα ε, να εμποδίζουν τους ε, νέους να έρθουν στη χώρα και να ακολουθήσουν τη σωστή κατεύθυνση και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται. Ευχαριστούμε η κυρία Αρνόβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, μέσα στην έκθεση αυτή βλέπουμε τρεις βασικές, τρία βασικά στοιχεία αν θέλετε. Η πρώτη ε, λέξη κλειδί είναι εκπαίδευση κάτι πολύ σημαντικό από τα πρώτα χρόνια της ζωής, ε, από την προσχολική ηλικία. Εκεί αρχίζουμε να προωθούμε τις βασικές ε, δεξιότητες ε, στους νέους. Στη συνέχεια η δεύτερη λέξη κλειδί είναι η ψηφιοποίηση. Ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες βοηθούν τους νέους να καταλάβουν και τις ανάγκες των επιχειρηματιών. Και τρίτη λέξη κλειδί επιχειρήσεις. Ε, οι επιχειρήσεις που με τη τεχνογνωσία τους μπορούν να βοηθήσουν τους νέους ε, στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να είναι τμήμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε. Έτσι ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ομιλητών και ακούμε τώρα τον Επίτροπο για να απαντήσει. Επίτροπος Ναυραζίτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Σόιντροβα την συγκήτριά μας είναι πάρα πολύ ε, καλή η έκθεσή της και περιέχει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις αυξημένης βαρύτητας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε αυτό το ζήτημα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι πλέον ε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ρημότητα ε, που μας επιτρέπει να σημειώσουμε συγκεκριμένη πρόοδο. Δεν μπορούμε πλέον να αναρωτιόμαστε αν, θα, ε, μπορεί, αν μπορεί να διδαχθεί η επιχειρηματικότητα, αν ο σωστός χώρος είναι μία τάξη. Όχι, θα πρέπει να επικεντρωθούμε πλέον στο πώς θα διδάξουμε την επιχειρηματικότητα στα σχολεία και πώς θα έχουμε μια κρίσιμη μάζα ε, μαθητών και στη συνέχεια φοιτητών. Εκμάθηση της επιχειρηματικότητας. Τι σημαίνει, δεν είναι μόνο η σύσταση της επιχείρησης, όχι. Θα πρέπει η εκπαίδευση να επιτρέπει την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, αλλά και αξιών. Αυτό είναι ακόμη σημαντικότερο. Ε, ανάληψη πρωτοβουλίας σε δημιουργικότητα, ανθεκτικότητα, το να μαθαίνει κάποιος από τα λάθη του, ε, να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του μεταξύ άλλων δεξιοτήτων. Ε, εξακολουθούν να είναι απαραδεκτά υψηλά τα ποσοστά ανεργίας των νέων με την ε, διδαχή και την η ε, γενίκευση της επιχειρηματικότητας θα μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτή την έλλειψη αντιστοιχίας ανάμεσα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και την προσφορά των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε δε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ω ε, βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση του αποκλεισμού γιατί αυτό δεν είναι πλέον έκτημα μόνο μιας κοινωνικής τάξης. Ξαναλέω ότι έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα στο παρελθόν και οφείλουμε να αναγνωρίζουμε και την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 12 η Δεκεμβρίου 2014 βλέπουμε τι αναφέρεται για την επιχειρηματικότητα και αναφέρονται και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ε, εκπαίδευση και κατάρτιση στα σχολεία αλλά και τη διαβίω εκπαίδευση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από αυτές τις δράσεις. Πρώτον, και σημαντικότερο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ε, ε, που επιχειρεί την ενσωμάτωση ε, στη δακτέα ύλη των πανεπιστήμιων της επιχειρηματικότητας στις κοινότητες νέων τεχνολογιών και καινοτομίας. Παρακολουθούν μαθήματα επιχειρηματικότητας συμπληρωματικά ως προς την επιστημονική του κατάρτιση. Δεύτερον, η πρωτοβουλία για την επιχειρηματικότητα. Βάσει των στάσεων της έκθεση, θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώνει και να υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία που δρομολογήσαμε που κινούμε τον ΟΣΕ το 2013 για να υποστηρίξουμε την ανώτερη εκπαίδευση και να αναπτύξουμε νέα εργαλεία και καινοτόμους οργανισμούς για την πρόθεση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Σήμερα έχουμε περίπου 500 Ινστιτούτα Επιχειρηματικότητας και συνεχίζουν συνεχίζεται να αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων. Χάρη στο Εράσμους είναι 50.000 φοιτές, ένα στους πέντε είχαν ε, πρακτικές ασκήσεις επιχειρήσεις το 2013 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις συμμαχίες γνώσης, ε, δηλαδή προγράμματα συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, ε, πρόγραμμα ίδρυσης πολλών επιχειρήσεων σε 20 διαφορετικά σχολεία, σε 5 διαφορετικά κράτη-μέλη. Θα σταματήσω εδώ. Είναι μακρύς ο κατάλογος των δράσεων και δεν, ήρθα εδώ για να αναφερθώ σε αυτές τις δράσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά για να ε, εξερευνήσουμε ποιος είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον για να υποστηρίξουμε την διδασκαλία της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό φαίνεται στην έκθεση είναι δεξιότητες νέων τεχνολογιών της πληροφορίας. ICT, κέρια σημασία ε, στη σημερινή κοινωνία κυρίως για τους συνόρους. Πρέπει να βρούμε τρόπους, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρον αυτέ τι ευκαιρίες για του νέου επιχειρηματίε. Ε, δεύτερον, αναγνώριση των ε, δεξιοτήτων επιχειρηματικότητα, η αξιολόγηση και η πιστοποίησή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που, ε, κάτι που θα μου επιτρέψει και την κινητικότητά του είναι υψής τη σημασίας. Και πάλι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια κρίσιμη μάζα νέων επιχειρηματιών και να μεριμνήσουμε ούτω ώστε στα βιογραφικά σημειότητα να το όλο και περισσότερο ω τέτοιε οι δεξιότητε που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ε, και ε, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την διδασκαλία τη επιχειρηματικότητα ε, στα σχολεία και στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα θέλαμε τα επόμενα χρόνια να μεγενθύνουμε ακόμη περισσότερο αυτά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει σε συνεργασία με τους αρμοδίους επιτρόπους. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι άλλοι σημαντικότατοι κέριοι φορείς της οικονομίας στα κράτη-μέλη όπως οι επιχειρήσεις θα μας βοηθήσουν σε αυτό το ε, εγχείρημά μας. Ευχαριστούμε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται